take your seats as quickly and swiftly and quietly as possible. Παρακαλώ καθίστε με κάποια ησυχία. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. I also have a flight, so I'm, I'm doing the vote and then I'm off. Okay. If there are no objections, the agenda can be approved. Λοιπόν, μπορεί να γίνει δεκτή η ημερήσια διάταξη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, του ε, Σεπτεμβρίου δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα και αναβάλλεται η έγκριση για τον Νοέμβριο. Δυστυχώς καθυστερούν οι μεταφράσεις. Έχω ορισμένε τώρα ανακοινώσει. Οι αναφορές και η ΛΥΜΠΕ ασχολούμεθα με το θέμα του Ombudsman και της έκθεσής του για το Frontex, σύμφωνα με το άρθρο 55. Αυτό θα γίνει στην συνάντηση την κοινή που θα κάνουμε τον Νοέμβριο στις 10. Οι κυρίες κυρίες Κέλλερ και Μετσόλα θα παρουσιάσουν την πρότασή τους. Είναι μάλλον μια συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Στις 11 Νοεμβρίου τώρα, 12η μεσημβρινή είναι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών οι οποίες μπορεί να κατατεθούν μόνο στην Αγγλική και στις 12 θα συναντηθούν από κοινού οι Επίτροπες στην δική μας τακτική συνεδρίαση και στις 16 ακριβώς θα υπάρξει μια κοινή συνάντηση της ΛΥΜΠΕ και των αναφορών. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΛΥΜΠΕ, επαναλαμβάνω. Δεύτερον, ε, το εργαστήρι Γιούρι και Πέτησιο ε, θα διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 12.30 στις 9 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα σας διανεμηθεί σε εύθετο χρόνο. Έχω και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, στις οποίες θα επανέλθω αργότερα όμως. Τώρα, έχω κάποιες πρόσφατες ειδήσει γύρω από τη συνάντηση των συντονιστών, η οποία μόλις προηγήθηκε. Εμείς πήραμε κάποιες αποφάσεις για την ημερήσια διάταξη του μηνός Νοεμβρίου. Υπήρξαν κάποιες διαφορές, διαφοροποιήσεις. Υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία λοιπόν, όπως είπα για την έκθεση Frontex, με βάση την έκθεση του Ombudsman. Τροπολογίες όπως είπα θα κατατεθούν μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα χρησιμοποιηθεί η επιταχυν, ε, επιταχυνόμενη ουσιαστικά συγκεκριμένη περίπτωση διαδικασία. Υπάρχει επίσης ε, και η, η 1156 για την κυδαιμονία των παιδιών ε, τον Δεκέμβριο θα συζητηθεί. Τώρα οι αναφορές για τους λύκους θα συζητηθούν τον Νοέμβριο. Και οι αμφισβητούμενες συστάσεις υιοθετήθηκε η πρότασή μου με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Για δέκα αναφορές για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας έγινε ψηφοφορία μεμονωμένη για κάθε μία και ε, κηρύχθησαν απαράδεκτες και οι δέκα. Στη συνέχεια περάσαμε στην αναφορά 2076 παραμένει η αρχική σύσταση, θα παραμείνει ανοιχτή δηλαδή η αναφορά. Η 2213 για τις διακρίσεις στη Μάλτα. αποφασίσαμε ότι θα στείλουμε μια επιστολή στην Επιτροπή, θα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες και θα ενημερώσουμε και τις αρχές της Μάλτα για την τροπολογία 2214 για τις αποζημιώσεις της γερμανικές θεωρήθηκε παραδεκτή. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα στείλουμε την αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω έρευνα και ε, για ενημέρωση θα αποσταλεί ε, μια επιστολή στη γερμανική κυβέρνηση και στην ελληνική κυβέρνηση προς ενημέρωση. Η 0927 αναβάλλεται για την επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Δεν ξέρω τι άλλο έχω να σας πω εδώ. Λάβαμε υπόψη μας επίσης και το πρόγραμμα της ερευνητικής αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το τελικό πρόγραμμα θα το λάβετε σε λίγες μέρες όσοι εσείς τουλάχιστον συμμετέχετε στην αποστολή αυτή τη διερευνητική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Ε, σας ζητώ να βάλετε την κάρτα σας στη σχισμή. Με την κάρτα θα ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη γνωμοδότηση για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη, ανάγκη μιας ολοστικής νέας προσέγγισης στην μετανάστευση. Δεν υπάρχω. Συνοδοστική. Ένα. Υπέρ. Κατά. Να αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική δύο υπέρ. Κατά. Όχι. Αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές Ολίγες, αλλά εγκρίνεται. Τριάντα δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, συμβαστική τέσσερα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές απερίφθη. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά χες ρίπτε 43 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 44 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 46 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 55 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 56 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά χες εγκρίνεται Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Multitasking, multitasking. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αρχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, επαλήθευση, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τη συμβιβαστική 11. And the vote is closed. Έληξε. Εγκουρίνεται. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 91 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. χες απορρίπτεται. 93 επίσης σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Yes. Okay. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Yes. Απορρίπτεται. 96 υπέρ Α, όχι, όχι, σε δύο τμήματα είναι, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εσ. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. 97 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 99 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χες απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται έληξε Ο, εγκρίνεται, εγκρίνεται με τρεις αποχάς. Συγχαρητήρια τον Και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάρω την τελευταία πληθύση για τη Σουηδία και η Ρομπέρτα Μέτσολα υποσχέθηκε να συμπροεδρεύσει, αλλά δεν ήρθε, άρα, άρα, δεν είναι εδώ η Ρομπέρτα, Υποσχέθηκε ότι θα έρθει και δεν ήρθε. Είναι όμως ήρεμη συνεδρίαση χωρίς προβλήματα. Έρχεται μου λένε, έρχεται. Α, εντάξει, μία μικρή παύση λοιπόν. Σας εύχομαι καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Hello everybody. Let's move to the next item, item number 9. Συνεχίζουμε. Στο πρόγραμμα λοιπόν τη Επιτροπή. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκέριγκα. Είναι μαζί μας, θα της δώσω αμέσως το λόγο. Πριν όμως δώσω το λόγο ε, στους σκιώδεις στη συνέχεια. Έχετε το λόγο κυρία Γκέριγκερ. raportu prezentowałam już Państwu na poprzednim posiedzeniu, Κοιτάξτε, έχω παρουσιάσει τα βασικά επιχειρήματά μου. Τώρα έχω το σύνολο της έκθεσης, διαβάστε την, εκτιμήστε την και αν θέλετε καταθέστε και τροπολογίας. Σύντομα λοιπόν θα σας πω ότι πρόκειται για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών για το 2014. 2.714 αναφορές, μείωση κατά 6% δηλαδή σε σύγκριση με το 13. Οι αναφορές βέβαια σημαίνουν και πληροφόρηση για τον τρόπο εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και τις περιπτώσεις παραβιάσεων. Είναι πολύ σημαντικό για μας ως νομοθέτες. Θέλουμε λοιπόν η νομοθεσία που δημιουργούμε να είναι θετική για τους πολίτες αλλά και σεβαστή από αυτούς, από όλους, ανεξαρτήτως επίπεδου. 127 ε, Μπράβο udział w debatach Λοιπόν, ήρθαν πάρα πολλοί αναφέροντες ή αναφερόμενοι, 700 περίπου, αλλά δεν έγινε καμία αποστολή το 2014, γιατί ήταν έτος ευρωεκαλογών. Οι πολίτες πάντως λένε οι ίδιοι ότι τέτοιες αποστολές είναι θετικές αυτό που δεν τους αρέσει είναι ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες παρουσίασης περισσότερο των απόψεών τους προς τις τοπικές αρχές. Ή διστάζουν ή δεν έχουν χρόνο ή φοβούνται. Άρα θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή Αναφορών. Πολύ συχνά μαζί με τα παράπονα των αναφερόντων ή αναφερομένων στέλνουν αναφορές και στην Κομισιόν και ένα τρίτο αυτών αφορούν παραβιάσεις της νομοθεσίας από κράτη-μέλη. Για πολύ καιρό είχαμε τα ίδια θέματα και άρα πρόκειται για σπατάληση εδώ για θέματα όπως ελεύθερη διακίνηση, διαχείριση υδάτων κλπ. Τα ίδια θέματα επί χρόνια. Πέρυσι επίσης συγκεντρώθηκε η προσοχή μας στο θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών που είναι ένα νέο εργαλείο. γάναμε μια σειρά ακροάσεων και η πρώτη από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι έτοιμη για νομοθέτηση από την Κομισιόν. Πρόκειται για το δικαίωμα στο νερό. Άλλο πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία με τις τοπικές εθνικές αρχές για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου ανέφερα ήδη ότι συναντούμε άμεσα πολίτες και τους ανοίγουμε την πόρτα για να συζητήσουμε καθώς και τοπικές αρχές ε, και συζητούν με τις τοπικές αρχές και μέσω του, της Επιτροπής μας. Επίσης ε, οργανώνονται καμιά φορά πιο πρακτικής φύσης συνεδριάσεις που αφορούν τον συνδυασμό αναφορών με παρόμοια αιτήματα. Κάτι άλλο, ο σεβασμός του, της χάρτας των θεμελιωδών και ιδιαίτερα του άρθρου 51. Δυστυχώς αυτό δεν αφορά όλες τις χώρες μέλη, αλλά ακόμα και σε εκείνες που δέχονται, που ε, επικύρωσαν τη χάρτα, το άρθρο 51 το επικαλείται συχνά η Κομισιόν διότι λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν η Επιτροπή Αναφορών ε, έθεξε το θέμα. Θελήσαμε να απαντήσουμε ότι η χάρτα είναι ένα συνοπτικό εγγράφο και πρέπει η Κομισιόν το άρθρο 51 να το ερμηνεύει διαφορετικά για να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες. Άλλο σημαντικό βήμα προς καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες ήταν το άνοιγμα ενός νέου ηλεκτρονικού δρόμου ή πόρταλ για να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν πώς πάει η αναφορά αν έχει γίνει αποδεκτή και τα λοιπά. Το δίκτυο Solvit επίσης είναι μια καλή λύση. Πρέπει όμως νομίζουμε το Solvit να ενδυναμωθεί από την Κομισιόν. Αυτό αναμένουν οι πολίτες. Επίσης, είχαμε καλή συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον προηγούμενο και την Έμιλι Ράιλι. Και τώρα θα ήθελα να δείτε τα στατιστικά στοιχεία αν σας ενδιαφέρουν που είναι οι πηγές της έκθεσής μου. και όπου βλέπετε πόσο σοβαρά παίρνουν οι πολίτες την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η έκθεση βρίσκεται σε όλες τις γλώσσες, γι' αυτό θα σας συστήσω να την ε, δείξετε και στους ψηφοφόρους σας ώστε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Συμφωνούμε ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για όσα κάνουμε. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η Επιτροπή μας. Τώρα, ο Σκιώδης του ΕΛΚ πρώτος δεν είναι εδώ βέβαια ο κύριος Μπέκερ, αλλά υπάρχει αντικαταστάτης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Μπέκερ δεν μπορεί να παραστεί. Θα συνοψίσω λοιπόν τι θα ήθελε να πει. Θα συνοψίσω αυτά που έλεγε. Λοιπόν, είναι πολύ ικανοποιημένο από την έκθεση της ΑΝΑΦ ιδιαίτερα για την αποδοχή των νέων τεχνολογιών που πλησιάζουν εμάς με τους πολίτες και εξοικονομούν και χουρήματα. Επίσης χαίρεται γιατί η Επιτροπή μας ε, έχει όλο και μεγαλύτερη, παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Συνεργάζεται με όλο και περισσότερες άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου και είναι ευγνώμων για την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχουν σαφέστερες διαδικασίες και διορίες που επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτές και βελτιώνουν έτσι τον κύκλο ζωής των αναφορών. Αναφέρει και μένα και όσα είχα κάνει για την προηγούμενη έκθεση. Κάτι άλλο που τονίζει είναι ότι θα ήθελε οι συγητές να καθορίζουν οι ημερομηνίε για τις συναντήσεις των σκιωδών. Μα ήταν καλό να συνανοηθούμε γρήγορα. Αυτά είναι τα σχόλια του κύριου Έκερ. Και εγώ ήθελα να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα πριν δώσω το λόγο σε άλλους κοιόδης. 22 Οκτωβρίου λίγη διορία τροπολογιών και στην Επιτροπή μας η ψηφοφορία 3 Δεκεμβρίου. Και στην Ολομέλεια μάλλον τον Ιανουάριο αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Τώρα η κυρία Αλβιόλ της Γκουέ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την γραμματεία γιατί πράγματι η έκθεση αυτή προϋποθέτει μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά από πλευράς της. Αλλά είναι σημαντική και για την Επιτροπή μας. Αντικατοπτρίζει σωστά τις εργασίες της Επιτροπής μας για το 2014 και να υπογραμμίσουμε εδώ την ανάγκη που υπάρχει οι αρχές των κρατών μελών να δείξουν μεγαλύτερη επιθυμία συνεργασίας και με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και είναι πολύ σωστή η αναφορά την οποία σημειώνει η συγκεκριμένη έκθεση με την χάρτα, για την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα καταθέσουμε ορισμένες τροπολογίες οι οποίες θα έχουν σαν στόχο ε, το να μην ε, παρετηθούμε κατά κάποιο τρόπο στα πλαίσια μιας σχετικής ικανοποίησης από την προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη παρουσία της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής στις Ολομέλειες, να ακούγεται, να φαίνεται περισσότερο και μέσω των αναφορών. Έχουμε επίσης και κάποιες τροπολογίες οι οποίες έχουν σαν στόχο την αύξηση της διαφάνειας της εργασίας μας έτσι ώστε να παίρνουν απαντήσεις ταχύτερα οι αναφερόμενοι μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών όπως το νέο πόρταλ. Μεγαλύτερη διαφάνεια και στη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επίσης και καλύτερη ενημέρωση για τις επαφές μας με τα διάφορα κράτη-μέλη υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το μέσο παρέμβασης και συμμετοχής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε ποια είναι πραγματικά η δραστηριότητά μας. Θα πρέπει να εντείνουμε επίσης τις δυνατότητες των διερευνητικών αποστολών τις οποίες κάνουμε και να ζητήσουμε επίσης ε, να αναθεωρηθεί σε βάθος ο κανονισμός για την πρωτοβουλία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη οργανώσει μια σημαντική ακρόαση γύρω από το θέμα αυτό, ενίσχυση του προσωπικού της γραμματείας έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στην ε, αντιμετώπιση όλων αυτών των αναφορών Υπάρχουν πάρα πολλές ε, τέτοιες αναφορές ε, οι οποίες έχουν σχέση και με την επικαιρότητα όπως με το TTIP, όπως επίσης και με το θέμα των, ε, το μεταναστευτικό τον τελευταίο καιρό. Θα συνεργαστούμε λοιπόν έτσι ώστε η έκθεση αυτή να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο Νομίζω ότι η βασική πρόταση είναι η πρόταση η οποία δείχνει το πώς δουλέψαμε σωστά το 2014. Σας ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Άουκεν εκ μέρους των Η Γιούλια δεν μπορούσε να είναι εδώ και άρα θα εκφράσω εγώ τις θέση της ομάδας μας. Ευχαριστώ για την έκθεση, χρήσιμη πρέπει ταυτόχρονα να προσέξουμε να μην ε, ευλόγαμε υπερβολικά τα γένια μας γιατί έχουμε κάποια προβλήματα. Καταρχάς, το web portal. κατάσταση είναι τραγική, δεν, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς. Μας λένε άνθρωποι, μα δεν δουλεύει. Και νομίζω ότι αυτό ε, ε, πρέπει να το σημειώσουμε ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση ασφαλώς. Και επιτρέψτε μου που θα εστιαστώ μόνο σε αυτά που έχουμε να επικρίνουμε. Όταν μιλούμε για το τρόπο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθυστερεί πολύ πολλές φορές και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο εαυτούς ή τον αναφερόμενο για το φόρτο εργασίας. δουλειά μας είναι να μιλήσουμε ξεκάθαρα και σε αυτό. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και κύρια παρατήρηση. Χάνουμε λίγο το, το κέντρο της προσοχής μας ως προς τον πολίτη. Δηλαδή κηρύττουμε παράδεκτες ε, αναφορές, είχαμε παράδοξες βέβαια εμπειρίες πριν από μια ώρα που συζητούσαμε για το πώς χειριζόμαστε τα θέματα αυτά μεταξύ μας. Πολιτική είναι η αναφορά, η υπόθηκε, την ψηφίζουμε, δεν την ψηφίζουμε. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και να βοηθήσουμε να προχωρούν οι αναφορές για το καλό των πολιτών, για να βλέπουν απαντήσεις στις ε, υποθέσεις τους χρειαζόμαστε πιο, πολλές, ε, πιο πολλούς πόρους στη γραμματεία για να είμαστε αποτελεσματικοί και όχι απλώς να ξεφορτωνόμαστε τον πολίτη, γιατί μερικές φορές φαίνεται αυτό να επιδιώκουμε μόνο. Και να είναι αυτό μόνο, το μόνο μας κατόρθωμα. Ας ε, εστιαζόμαστε λοιπόν περισσότερο στις ανάγκες ε, και στις αναφορές. Αυτό έτσι ώστε να μπορεί και η γραμματεία μας να κάνει εις βάθος δουλειά στις διάφορες υποθέσεις. Και επίσης. Για το για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση. Για το TTIP ακούστηκε ότι υπάρχουν ας πούμε εκατομμύρια υπογραφές. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πρωτοβουλία πολιτών αλλά διαμαρτυρία. Αλλά και σε αυτό έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε περιγράψει σωστά τι σημαίνει ε, έτοιμα ή αναφορά πρέπει να του εξηγήσουμε περί τίνο πρόκειται για να καταλάβουν ότι δεν τους ε, πετάμε έξω, αλλά ότι χρειάζεται να βρουν έναν άλλο τρόπο να διαχειριστούν το, τη διεκδίκησή τους. Την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, επί παραδείγματι, πολιτών. Ή ότι εμείς είμαστε ο τρόπος να επικοινωνήσει ο πολίτη με, με το κοινοβούλιο πιο άμεσα. Αυτό έχω κυρίως να σημειώσω. Και θέλω να το σημειώσω αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε σε κριτήριο ε, την πραγματική δουλειά και όχι το ότι ξεφορτωθήκαμε τους πολίτες. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Έφη. Και μετά ο κύριος, ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Αυτή η ετήσια έκθεση είναι ιδιαίτερως χρήσιμη για την αξιολόγηση της εργασίας αυτής της Επιτροπής η οποία έχει άμεση σχέση με τον πολίτη. Βρίσκουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστούν και θα σημειωθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα υποστηρίξω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Όλες αυτές είναι παρατηρήσεις ιδιαίτερα σωστές, διευκολύνουν τις εργασίες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σταθώ στο θέμα ε, θέμα του, του, της πρωτοβουλίας για τους πολίτες, ε, διότι η πρωτοβουλία των πολιτών δεν είναι κάτι το οποίο έχει αυτή τη στιγμή να δώσει τις δυνατότητες στους πολίτες, αυτές τουλάχιστον που χρειάζονται. Και η χρήση του μέχρι τώρα ήταν σχετικά απογοητευτική. Ενώ εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει αναθεώρηση του συγκεκριμένου μέτρου έτσι ώστε οι πολίτες να βρουν τρόπους και μέσω της πρωτοβουλίας των πολιτών να συμμετέχουν στην διακυβέρνηση της Ένωσης. Και η διαφάνεια φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, όπως έχουμε ήδη πει, όπως έχουμε ήδη προτείνει. Το πόρταλ το οποίο έχουμε θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλα τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ε, υποτίθεται κάποιες τεχνικές δυσκολίες σε σχέση ε, με, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο τεχνικό και όλοι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, το πόρταλ αυτό με μεγάλη ταχύτητα και να ανταποκρινόμεθα έτσι με πιο αποτελεσματικό τρόπο στα αιτήματα των ε, πολιτών. Πάντως να συγχαρώ ακόμα μία φορά την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Ε, καλύτερη λειτουργία της ε, Επιτροπής μας και βεβαίως θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Υπάρχουν ορισμένα θέματα σημαντικά τα οποία αναδείχθηκαν. Πρώτα απ' όλα είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή μας δέχεται πάρα πολλά αιτήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδοκούν, αναμένουν την δράση της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να έχουμε την επίλυση σημαντικών προβλημάτων τους. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό διότι δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα. Το ζήτημα όμως είναι ότι μια επιτροπή σαν τη δικιά μας πρέπει να έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα αυξημένα αιτήματα. Επομένως πρέπει να οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου ε, πράγματι αυτό να, μπορεί να συμβεί. Ε, άρα χρειάζεται συγκεκριμένη τεχνική υποδομή, χρειάζεται στήριξη από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και όμως δεν το έχουμε. Το δεύτερο θέμα που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή ε, έχει άμεση σχέση και ε, αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Μια σημαντική ρήτρα που υπάρχει στην συνθήκη, σύμφωνα με την οποία ε, εάν υπάρξουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές από συγκεκριμένο αριθμό κρατών και αυτές είναι από τους πολίτες, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη υποχρέωση της Επιτροπής της Κομισιόν να προχωρήσει σε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Ήδη δεν έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια. Γίνονται επίσης ενέργειες και από την πλευρά της Κομισιόν λίγο να περιοριστούν οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ίδιων των πολιτών. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ και να βγάλουμε συμπεράσματα, ώστε να διευκολύνουμε πραγματικά την άσκηση της πρωτοβουλίας πολιτών ένα δημοκρατικό δικαίωμα των ίδιων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αντιμετωπίζουμε βεβαίως και είδαμε νομίζω σωστά θέματα σημαντικά όπως είναι το ζήτημα της ε, μετανάστευσης, ε, το προσφυγικό και νομίζω σε αυτό και εκθέσεις συντάσσουμε αλλά και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις για να συμβάλλουμε να αντιμετωπιστεί αυτά τα θέματα που είναι ε, σύγχρονα και ιδιαίτερα σημαντικά θα έλεγα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως για τους πολίτες, για τους ανθρώπους που ε, καταδιώκονται από διάφορες εμπόλεμες ζώνες και έρχονται στην Ευρώπη να σωθούν. Και φυσικά ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι το θέμα της TTIP, μας έχει αποσχολήσει, βλέπουμε μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3 εκατομμύρια υπογραφές για το ζήτημα αυτό, επομένως η Επιτροπή μας πρέπει να το δει, διότι εμείς είμαστε η Επιτροπή που πραγματικά συνδέεται με τους ίδιους πολίτες. Άρα λοιπόν αυτό σε σχέση επίσης και με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που πρέπει να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ότι πρέπει να καταλάβουν τα κράτη ότι κάποτε πρέπει να εφαρμόζουν την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ότι θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο συνεργάσιμη και λειτουργική με εμά η ίδια η Επιτροπή. Νομίζω είναι συμπεράσματα τα οποία όλοι έχουμε βγάλει. Θα τα παρουσιάσουμε και αργότερα, θα κάνουμε και τροπολογίες για να συμβάλλουμε να έχουμε μια θετικότατη έκθεση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε άλλο κύκλο όταν θα ξανασυζητήσουμε και θα έχουν κατατεθεί και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you very, very much. Um, I'll give the floor now to any other members who would like Σας κατευχαριστούμε. Όποιος άλλος θέλει το λόγο. Μορμπάτη. Μαζί. Ναι, σύντομα, σύντομα. Συμφωνώ με ό,τι είπαν οι συνάδελφοι, αλλά σκέφτομαι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Ερωτώ λοιπόν τον εισηγητή 124 αναφορές είπατε. Πόσες αφορούσαν ε, παράβαση. Γιατί εδώ ακούμε και για αναφορές ε, όπου αν δεν αποδείξουμε ότι μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα στο κράτος μέλος τίθεται το ερώτημα σε... Ε, γιατί σε τι χρησιμεύει επί 124 αναφορών πόσες παραβιάσεις τι έγινε γιατί όσο πιο πολύ δείξουμε ότι η Επιτροπή μας μπορεί πράγματι να παίξει ένα ρόλο και για την πληροφόρηση γιατί πολλές φορές οι πολίτες δεν έχουν τις πληροφορίες και γίνεται παραβίαση των οδηγιών τόσο πολύ μπορούμε να, περισσότερο μπορούμε να δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και οι πολίτες θα πούνε, α, να, να η αποτελεσματικότης. Και έτσι θα αναγνωριστεί η Επιτροπή μας. Αλλά βέβαια αυτό απαιτεί και κυρώσεις. με κυρώσεις, αλλιώς δεν αρκεί. Ευχαριστούμε πολύ τώρα ο της Επιτροπής της Κομισιόν, ο κ. Λεαρντίνη και μετά η κυρία Γκέριγκερ για να καταλήξει σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω. Η Κομισιόν ε, δέχεται αυτή την έκθεση ασμένος και γιατί αναγνωρίζει ότι είμαστε συνέτεροι σε αυτήν, εταίροι σε αυτήν την επιχείρηση. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Επιτροπή σας πριν από ένα χρόνο, είχατε ήδη συζητήσει το θέμα των καθυστερήσεων που είχαν σημειωθεί ε, με τα χρόνια και νομίζω ότι από τότε έχετε προοδεύσει πολύ. Καθάρισαν τα πράγματα. Κατ' εμάς, ε, το κατά πόσον μία αναφορά είναι αποδεκτή ή όχι δεν είναι θέμα άσπρου μαύρου ούτε καθαρά ο αριθμός των αναφορών. Το θέμα είναι αν γίνεται λύση στα προβλήματα. Ας πούμε εναλλακτική λύση διενέξεων διαφορών και αν είναι αυτός ο καλύτερος δυνατός τρόπος για τους πολίτες για να λύσουν το πρόβλημά τους. Τότε να το χρησιμοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα διαχείρισης των αναφορών διεκπαιρέωσης. Εκεί παραπονούν ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος για να απαντήσει η Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να σας τονίσω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είμαστε οι μόνοι παράγοντες. Πολλές φορές πρέπει να απαντήσουν και τα κράτη-μέλη και εκείνα είναι που καθυστερούν. Υπάρχουν θέματα μετάφρασης και πάνω απ' όλα όμως είναι το θέμα του αν απαντούν εν καιρό στα κράτη-μέλη στα αιτήματα που τους στέλνουμε. Γι' αυτό χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρόσκληση που κάνετε σε εκπροσώπους των χωρών μελών στις συνεδριάσεις σας για να ακούσετε από πρώτο χέρι τα πράγματα χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να περνάτε από την Κομισιόν. Τρίτον, η ανάγκη να τηρούνται ενήμεροι οι αναφέροντες. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο δυνατόν συχνότερα ανακοινώσεις τύπου όποτε γίνονται γνωστές παραβιάσεις και φυσικά αν μας το ζητήσετε μπορούμε να έρθουμε να εξηγήσουμε που ακριβώς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επί παραλήψη. Τέλος για το 51 της χάρτας. Εδώ πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν υπάρχει ευρύτερη ή στενότερη ερμηνεία των δικαιωμάτων. Το 51 προβλέπει ότι η χάρτα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη μόνον όσταν και στο βαθμό που εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Συμφωνώ ότι υπάρχουν όρια για την εφαρμογή της χάρτας, αλλά μόνο στο βαθμό που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη το ενωσιακό δίκαιο μπορούμε να κάνουμε κάτι και αυτό βέβαια το κάνουμε όταν υπάρχουν οι λόγοι, όταν συντρέχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκέριγκερ τώρα για να απαντήσει σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ χρήσιμη συζήτηση. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Και τώρα θα αναφερθώ στις παρατηρήσεις σας. για το πόρταλ. Δεν λειτουργεί τέλεια. Ναι, προφανώς, το δέχομαι. Δεν έχουμε φτάσει που θα θέλαμε να είμαστε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση όμως. Μία επιτυχία είναι ότι περνούσε πολλής χρόνο έω και χρόνια για να ε, επεξεργαστούμε μία αναφορά. Τώρα βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει κλείσει. Και βεβαίως βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πόρταλ ε, για να υποβάλλονται οι αναφορές χωρίς δυσκολίες. Αυτό όμως δεν εξαρτάται πάντα από μας. συμφωνώ δε ότι χρειαζόμαστε επιπλέον προσωπικό στη γραμματεία. Αυτό όμω πώς συνάδει με τη στρατηγική για οικονομίες. Γιατί ξέρετε είμαι και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Και ξέρω ότι μειώνονται μάλλον οι θέσεις εργασίας, δεν αυξάνονται. Άρα και εγώ θα ήθελα περισσότερη αποτελεσματικότητα στις εργασίες, αλλά πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Είναι μια επιθυμία η οποία όμως θα μείνει ελπίδα φρούδα διότι δεν μπορεί να στηριχθεί σε πραγματικές λύσεις. Και κάτι ακόμη. Στην Επιτροπή μας ποτέ για να απαντήσω στο σχόλιο των πρασινών. Δεν προσπαθήσαμε να απαλλαγούμε από μια αναφορά. Όχι, δεν ξεφορτωνόμαστε. Ούτε πιστεύω ότι θέλουν, ότι αντιλαμβάνονται οι ε, πολίτες ότι δεν τους λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά δεν πρέπει και να ξεπερνούμε το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Εάν δεν έχουμε αρμοδιότητες, δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις τέτοιου τύπου. Και συμφωνώ από την άλλη ότι δεν είναι δυνατόν να ε, αφήνουμε ένα θέμα και απλώς να το κλείνουμε. Πρέπει να ε, βρούμε έναν τρόπο να μην απαντούμε μόνο αρνητικά στον αναφερόμενο αν πρόκειται για ζήτημα αρμοδιοτήτων, αλλά να βρίσκουμε μία λύση. Ακόμα και αν πρόκειται για ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Μπορούμε παραδείγματι να στέλνουμε στις εθνικές αρχές ε, μια αναφορά και να ζητούμε να το, να αντιμετωπίσουν το θέμα. Μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Άρα μπορούμε να βελτιώσουμε και την επικοινωνία μας με τα εθνικά κοινοβούλια Φερρυπίν. Και να τα αξιοποιήσουμε και εκείνα ως ε, σύνδεσμο. Για να μην νομίζει και ο αναφερόμενος ότι άπαξ και κρίθηκε αναφερο, απαράδεκτη μία ε, προσφυγή του δεν υπάρχει τρόπος να επιληθεί, να αντιμετωπιστεί. Έχουμε λοιπόν τώρα τις απαντήσεις της Επιτροπής, εξηγήσεις των κρατών μελών. Πρέπει να κοιτάμε τις εξετάσεις ε, και από τη νομική προοπτική των εθνικών ε, νομοθεσιών, να κοιτάμε δηλαδή αν μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε στο να αντιμετωπίσει σε εθνικό επίπεδο μια υπόθεση και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι οι δραστηριότητες μας, και αυτό το επιβεβαιώνει και η Επιτροπή, η δουλειά μας είναι να εξηγούμε μένα, αλλά ίσως δεν ε, κοιτάμε πάντα εάν έχουν αξιοποιηθεί μέσα που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Γιατί δεν είστε παιδί των αυτό. Σε αυτό λοιπόν περιμένω περισσότερα σχόλια αγαπητοί συνάδελφοι. Από ό,τι βλέπω στα αγγλικά μόνο το έχουμε προς το παρόν. Δεν ξέρω αν η διαδικασία είναι τύπου fast track. Και αν υπάρχει τρόπος να ετοιμάσουμε τις τροπολογίες και σε άλλες γλώσσε, να τις δούμε και σε άλλες γλώσσε. Ή δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, ή δάλος μόνο στα αγγλικά. Θέλω να θυμάστε ότι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το μεσημέρι έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε τις προτάσεις σας και παρακαλώ τη γραμματεία να μας πει αν έχουμε αυτή τη δέσμευση με τα αγγλικά μόνο ή όχι. Ναι, ρώτησα τη γραμματεία και μου λένε ότι μπορείτε να καταθέσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα, όχι μόνο στα αγγλικά. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Έτσι λοιπόν, περνάω στα αγγλικά. Σημείο 10. Ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Διαμεσολαβήτριας 2014. έκθεση Ρέιλι αρχικά για ολόκληρο το έτος. Την είδαμε την έκθεση της κυρίας Ρέιλι τον Ιούνιο και μετά ανέλαβε η κυρία Καβεσόν την οποία και παρακαλώ να παρουσιάσει την έκθεσή της για να δώσω στη συνέχεια το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Επειδή έχουμε μεγάλη ε, καθυστέρηση στο πρόγραμμά μας. Σας παρακαλώ όσο δυνατόν πιο σύντομα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, βεβαίως θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη κατά το δυνατόν. Πράγμα που δεν είναι πολύ εύκολο. Τέλος πάντων. Είναι η πρώτη έκθεση της καινούργιας διαμεσολαβητρίας και προσπαθεί να ιεραρχήσει τις πρωτοτεραιότητες της θέσης της κλπ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω από την αρχή ότι η έκθεση της διαμεσολαβητρίας μου φαίνεται καλή. Καλή. Ενισχύει τη διαφάνεια στα θεσμικά όργανα αυξάνει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και δίδει εγγυήσει για τον σεβασμό γενικότερα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία κατέληξαν στο γραφείο του διαμεσολαβητή. Η μεγάλη πλειοψηφία πήγε εκεί μέσω του διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο αυτό είναι κατάλληλο και το ποσοστό αυτό αυξάνεται κάθε χρόνο. Ένα μέσο ιδιαίτερα ευέλικτο το οποίο χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Άνω των 2.000 λοιπόν απαντήσεων οι οποίες δόθηκαν με συγκεκριμένες συστάσεις, παραπομπές, Συγκεκριμένα υπήρξε και πιο επιμέρους ανάλυση 325 υποθέσεων. Είναι θετικά τα αποτελέσματα αυτά γιατί φαίνεται ότι χρησιμοποιείται η δυνατότητα την οποία έχει το γραφείο του Ομπούτσμαν του διαμεσολαβητή να ερευνήσει κάπως τα πράγματα όταν αυτό παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον για τους πολίτες. Λοιπόν, είναι μια καλή έκθεση, είναι μια καλή αρχή στην εντολή της διαμεσολαβήτριας στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι η πρώτη της περίοδος. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η διαφάνεια μέσα στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η διαμεσολαβήτρια είναι κάτι το οποίο απαιτεί ο Ευρωπαίος πολίτης. Γενικά η υπηρεσία αυτή του διαμεσολαβητή γενικά έχει προωθήσει διάφορες μορφές εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πολιτών, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα των εργασιών της. Είναι θετικές οι δημοσιεύσεις αυτές. Είναι σαφής η ταξινόμηση επίσης των στοιχείων που δημοσιεύονται και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προς τις ε, οι αλληλογραφίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις Ιρλανδικές Αρχές κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Υπάρχει το θέμα της δημοσίευσης της προόδου των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία TTIP. Όλα αυτά είναι μικρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι ε, έχει προχωρήσει η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας πάρα πολύ σημαντικής την οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί της είναι σημαντική και η ανάλυση η οποία έχει γίνει από πλευρά της υπηρεσίας αυτής και από πλευρά των κοινοτικών αρχών στα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες όπως ο τομέας της υγείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και σε άλλες περιπτώσεις όπως σαν παράδειγμα στα πλαίσια του καθορισμού του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Υπάρχει επίσης και το θέμα των κριτηρίων σχετικά με τη συμπερίληψη της διάστασης των φύλων. Είναι σημαντικό λοιπόν η υπηρεσία αυτή να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, να βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε τομείς ε, επίσης τους οποίους μπορεί η παρέμβασή της να είναι θετική όπως ε, η, ε, τα σχόλια τα οποία κάνει γύρω από τα θέματα της διαφάνειας της αγοράς των φαρμάκων έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις δοκιμές τις κλινικές που προηγούνται της κυκλοφορίας ενός φαρμάκου και για την επίτευξη μιας τιμολόγησης η οποία να ανταποκρίνεται και στο κόστος της έρευνας, της φαρμακοβιομηχανίας αλλά και του καινοτόμου των συγκεκριμένων φαρμάκων. Ε, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπόν, η ανάλυση την οποία κάνει της πολιτικής ε, ε, ε συνοχής, το πως ε, θέτει τα προβλήματα της κοινωνικής συνοχής, του πρόβλημα της φτώχειας, είναι απαραίτητο να υπάρξει βελτίωση και να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία και μεγαλύτερη τεκμηρίωση έτσι ώστε να εγγυηθούμε μεγαλύτερη, μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας. Υπάρχει επίσης και το θέμα των επαναπροωθήσεων και της σωστής λειτουργίας του Frontex ενός μηχανισμού ο οποίος πρέπει να εξυπηρετήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι ώστε το σύστημα αυτό να λειτουργεί με πιο ικανοποιητικό ε, τρόπο. Ε, προχωρεί επίσης και σε περαιτέρω άλλες αναλύσεις γύρω από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια των μεταναστευτικών φαινομένων που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό. Η ανάλυση η οποία επίσης έχει προστατηθεί για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών είναι προτάσεις σημαντικές και χρήσιμες και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. επίσης σημαντικά αυτά τα οποία λέγονται και για τους συμπολίτες μας με προβλήματα αναπηρίας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Ναι, ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Βαλέντς, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της και την επιμέλεια που έδειξε σε αυτήν την ναι. έκθεση. Η οποία δείχνει βεβαίω τη πραγματική ποιότητα της δουλειά της κυρίας Ουράιλη. Θα θυμάστε ίσω ότι από την αρχή που ανέλαβε τα καθήκοντά τη, επιδιώκει να διαφυλάξει τις βέλτιστε προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια διάλογο με τους πολίτες. Και πάνω απ' όλα θέλει να διαφυλάξει τη σχέση εμπιστοσύνη με τον, ε, μεταξύ πολίτη και ευρωπαϊκής δημόσιας, υπηρεσία. υπηρεσίας. Είναι καλή λοιπόν ισορροπημένη η έκθεση. Για να προσθέσω όμως κάτι και θα το συζητήσουμε βεβαίως με την εισηγήτρια και τους σχεδόν ίσως μπορούμε να επεκτείνουμε κάπως το πεδίο της εκθέσεως προκειμένου να καταγράψει την ε, σημασία της δουλειάς της Ομπούτσμαν στην διαφύλαξη του έργου του Ομπούτσμαν. έτσι ώστε να δείξουμε ότι η διαφάνεια στη δουλειά της ε, ο ορίζον 2020 κτλ ε, έχουν τη σημασία τους. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε μέσα από τις ε, συναντήσεις μας με τους κοιόδης και την συγκεκριά να το αναπτύξουμε περισσότερο για να επεκτείνουμε το φάσμα της ε, ε, εκθέσεως. Ωραία. Τώρα ο κύριος Μαριάς. Η εισηγήτρια παρουσίασε μια, ένα σημαντικό έργο και νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να στηριχτούμε για να συμβάλλουμε και εμείς με τις απόψεις μας ε, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη έκθεση σε σχέση με τη λειτουργία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για την ακρίβεια. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είχα θέσει και πέρυσι ε, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο ζήτημα αφορά τη διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι μια βασική αρχή που πρέπει να διακατέχει την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό βεβαίως ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την ε, ε, Κομισιόν, κυρίως όμως για την Κομισιόν. Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε διότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια τουλάχιστον ε, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων διεθνών συνθήκων και ειδικότερα στη διαπραγμάτευση της TTIP. Γίνονται μια σειρά πράγματα σε κλειστές πόρτες. Ε, δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση αυτή της σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία γίνεται ε, και στο τέλος θα κληθεί ευσπεσμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα κράτη να υπερψηφίσουν ε, ή να μην ψηφίσουν μια διεθνή σύμβαση. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει το θέμα της διαφάνειας της διαπραγματεύσεις διεθνών συνθηκών να αντιμετωπιστεί και είναι αντικείμενο της ίδιας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και από ό,τι ξέρω έχει κάνει και σχετικές παρατηρήσεις ήδη στην Κομισιόν η οποία προσπαθεί να δείξει δείγματα διαφάνειας. Το να μας λένε ότι ως Ευρωβουλευτές ε, στο πλαίσιο της TTIP μπορούμε να λάβουμε γνώση ορισμένων εγγράφων αλλά θα πρέπει να πάμε σε ένα ειδικό χώρο, να τα διαβάσουμε να μην μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις, να μην έχουμε κινητό μαζί μας, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι κάτι το οποίο ε, αντίκειται στην έννοια της διαφάνειας, του δημοκρατικού ελέγχου και της ε, συμμετοχής των ίδιων των ε, Ευρωβουλευτών. Το δεύτερο θέμα που είχα θέσει πέρυσι και νομίζω ότι φέτος ξανά έρχεται είναι η σύγκρουση συμφερόντων η οποία υπάρχει πολλές φορές σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει στο πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι υποτίθεται ανεξάρτητη νομισματική αρχή, να εποπτεύει το 80% των τραπεζών μάλλον τις συστημικές τράπεζες στην Ευρώπη που καλύπτουν το 80% των διαθεσίμων, να είναι μέλος της Τρόικας και να είναι και επιστοτής, δανειστής δηλαδή της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας έχοντας αγοράσει ομόλογα. Α, κάτι πρέπει να γίνει και αυτό είναι, πρέπει να το επισημάνουμε. Πέρυσι είχα καταθέσει μια τροπολογία που ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε από 200 συναδέλφους <laughs> αλλά καταψηφίστηκε από περίπου 400 συναδέλφους ε, στο, στο ζήτημα του ελέγχου της ε, σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της ε, λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ποιος θα είναι ο ρόλος του, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στο θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ σοβαρά. Πιστεύω βέβαια ότι υπάρχουν και θέματα διαφάνειας και στην ίδια τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ως διοίκηση, ως διοικητικός μηχανισμός, όχι ως πολιτική δράση, ελέγχεται και από τον ίδιο το διαμεσολαβητή. Άρα λοιπόν ε, θεωρώ ότι η έκθεση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, θα κάνουμε τροπολογίες για να επισημάνουμε και αυτά τα θέματα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάουκεν εξ ονόματος των Παρασίνων. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ και το Μεσολαβήτρια και την εισηγήτρια. Να έχω και εγώ καλή συνεργασία μαζί της. Εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες, την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισλανδία δεν υπήρχαν παλιά ombudsmen. Τώρα βέβαια υπάρχουν, ε, αλλά στις χώρες που ανέφερα ήταν πιο πολιτική η λειτουργία τους. In the old member states are ah, a little bit offended when the ombudsman... Όταν ο Ombudsman ασκεί κριτική βέβαια, οι περισσότεροι θίγονται. αλλά είναι καθήκον του ομπούτσμαν ή της ομπούτσγουμαν να το κάνει. Και πρέπει όλα αυτά που παίρνει υπόψη της στη δουλειά της να μας χαροποιούν. Να ενδυναμώσουμε αυτόν τον θεσμό της ομπουτσμανοσύνης διότι και οι εθνικοί ομπουτσμέν πρέπει να γίνουν πραγματικά ανεξάρτητοι. Μερικοί από τους υποψηφίους είχαν πει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι όπως οι επίτροποι. Μα τι λέτε τώρα, οι επίτροπη; είναι πολιτικός ορισμένη ή διορισμένοι ενώ ο Ομποτσμάν πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητος σαν δικαστής όχι σαν επίτροπος σαν δικαστής και θα ήθελα στην έκθεση να λέει δύο πράγματα πρώτον να ζητήσουμε πραγματική ρύθμιση για την καλή νομοθεσία ε, ε, ε, security around Καλή διοίκηση, καλή διαχείριση, καλή νομοθεσία. Αυτά θέλουμε. όχι να γίνονται πράγματα κατά των πολιτών. Άκουσα να λέγονται πολλά για διαφάνεια, αλλά έλεγαν οι άνθρωποι της Κομισιόν, ε, αν κάνουμε λάθος και αυτό φάνει, τι θα γίνει. Χωρίς λάθη δεν γίνεται τίποτα. Όχι. Όχι, όχι. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεύτερον, η... τα διαπλεκόμενα συμφέροντα ή οι διαμάχες συμφερόντων συμβαίνουν σε τόσο πολλά μέρη. Ξέρω ότι κυρία Οράλη το παλεύει, αλλά πολλοί θεσμοί το μπερδεύουν αυτό με την απλή διαφάνεια. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαμάχη συμφέροντος σε τέτοιες θέσεις. Καμία. τουλάχιστον για όσους παίρνουν αποφάσεις στο όνομά μας. Καθόλου καμία. Αυτές οι δηλώσεις που ζητάμε σημαίνει ότι δεν θα κάτσουμε και να δούμε αν είναι και πιστοί στις συζύγους τους και τέτοια. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. δεν θέλουμε αντιπλεκόμενα ή διαπλεκόμενα συμφέροντα. Αυτό είναι όλο. Αυτό ζητάμε. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των πολιτών κατά των αρχών. Μάλιστα. Η κυρία Εύη τώρα από την ομάδα της και παρακαλώ να είναι συγκεκριμένη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η κυρία Άουκεν, αλλά να ευχαριστήσω εδώ και την συνάδελφο Καμπεσόν. Η έκθεση αυτή νομίζω αντικατοπτρίζει με σωστό τρόπο το πόσο δύσκολη είναι η δουλειά ε, της διαμεσολαβήτριας. Θα ήθελα σε ένα σημείο να σταθώ λίγο. Το θέμα της πρόσβασης σε έγγραφα και σε πληροφορίες, όπως είπε και η ίδια. Το 30% των καταγγελιών αφορούν θέματα πρόσβασης σε έγγραφα και διαφάνειας. Αυτό το οποίο βιώνουμε πρόσφατα είναι η πρόσβαση για το έργο σύνδεσης ε, ε, το Ρήνο Λιών Σιδηροδρομικής Σύνδεσης Εκεί υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και μια μυστικότητα σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν ήδη γίνει και στις χρηματοδοτήσεις ε, για το μέλλον. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς ε, χρησιμοποίησαμε και τον κανονισμό 1049 του 2001 που προβλέπει την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούνται πάρα πολλές εξαιρέσεις και αποκλήσεις επιτρεπόμενες για να περιορίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση. Παρακάμπτεται ουσιαστικά η ενημέρωση και δεν επιτρέπεται ε, προς τους πολίτες και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ούτε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε για δίποτε μορφή πρόσβασης. Θα προτείνουμε λοιπόν κάποιες επιπλέον τροπολογίες εδώ, αλλά σε ένα έγγραφο το οποίο είναι πραγματικά ήδη πολύ πλήρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε το θέμα κυρία Καμπεσόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, παρατηρήσεις οι οποίες ήσαν ιδιαίτερα επικοδομητικές και τις οποίες θα λάβω υπόψη μου. Θα λάβω υπόψη μου λοιπόν τις συνεισφορές του καθενός και κάθε από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Λάιτεμ νούμερο Τώρα θα περάσουμε στο 11. 11. Ο αναφέρον πρέπει να φύγει στις 6 και γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομοι όλοι. Έχουμε δύο μάλιστα αναφορές, δύο. Η μία είναι της Μονίκ Τουζό και της Ντανιέλ Κενσόν. Εξ ονόματος του Collective pour les Realisations Ecologiques 06 και τον Μαρί Λούζ Ερνάντες Νικάζη και Αναμπέλα Γέγκερ για την περιβαλλοντική κατάσταση Παιδιάδα Βάρ Γαλλία και άλλη αναφορά για το ίδιο αυτό το τμήμα της Γαλλίας του Σεμπαστιάν Βαλαμπουά. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μονίκ Τουζό για πέντε ολόκληρα λεπτά. Is the petitioner in the room? Είναι στην αίθουσα η αναφέρουσα ή αναφερόμενη. Okay. Α, ναι, τότε καλά. Please keep to the time. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο Είμαι η κυρία Τουζό. Εμείς διαμαρτυρόμαστε για την ε, επιχείρηση εθνικού λέει συμφέροντος στην πεδιάδα του ΒΑΡ στο νότο της Γαλλίας. Η γεωγραφική κατάσταση σας παρουσιάζεται εδώ σε σύγκριση με την Νίκαια και την υπόλοιπη Γαλλία. 10.000 εκτάρια και 15 κοινότητες διαφορούνται εδώ. Είναι τεράστια επιχείρηση αλλαγής της χωροταξίας που κατ' πρέπει να τύχει αποτίμησης για τα και στις επιπτώσεις. Τον περασμένο Ιούλιο ένας δημόσιος οργανισμός που είχε αναλάβει τη διαχείριση ενέκρινε τον πρώτο του προϋπολογισμό ΠΠΑ, ΠΠΑ. και δεν έγινε καμία περιβαλλοντολογική αποτίμηση. Απαιτείται όμως. Οι διευθετήσεις να εξεταστούν στο σύνολό τους. εξόλου υπάρχει και ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Γι' αυτό προσεφήγαμε στο Διοικητικό Δικαστήριο της Νικαίας. Έχετε και αντίγραφο και θεωρούμε ότι εδώ πρόκειται για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Εδώ βλέπετε το κεντρικό τμήμα του ΒΑΡ με το πρόγραμμα BRIV. Με το πρόγραμμα που αφορά και τις δύο όχθες μάλλον του ποταμού. Εδώ προβλέπετε, όπως βλέπετε εκεί δεξιά, να μετακινηθεί ένα ορυχείο και πάνω απ' όλα όπως βλέπετε αριστερά υπάρχει και ένα πρόγραμμα μεταξύ God και Λαγκοστιέρο. Η God είναι μια κτηνοτροφική περιοχή και σε έκταση 25 εκταρίων προβλέπεται να επεκταθεί μέχρι το Λαγκοστιέρ. Θα ήθελα να σας πω ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνος πλημμυρών και υπάρχουν πολλές παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Εδώ είμαστε στο κάτω μέρος της κοιλάδας του Βάρ. Βλέπετε ότι στο κέντρο, εκεί που είναι άσπρη η παράσταση, φαίνεται ότι από την αρχή μέχρι τις εκβολές ε, θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα αυτό το πρόγραμμα του πεπερι και σας είπα ότι θα αυξηθούν οι κίνδυνοι των πλημμυρών και στη ζώνη αυτή προβλέπεται δόμηση παντού ακόμη και σε περιοχές που θα υποστούν τις πλημμύρες. Αριστερά βλέπετε γιατί η γη πρόκειται. Γη σφουγγάρι. Εκεί ακριβώς διάλεξαν να δομήσουν και δεξιά βλέπετε τι έγινε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015 η λάσπη εναποτέθηκε. Δεν υπήρξαν καταστροφές μόνο, και στις κάνε, μόνο στις Κάνες αλλά και εδώ. Ακριβώς γιατί οι γέες αυτές είναι σφουγγάρια. Εκεί απορροφάτε το νερό, το περισσεύον νερό. Εμείς θεωρούμε ότι εκεί ο καθένας μπορεί να καλλιεργήσει τα λαχανικά του και είναι σημαντικά όλα αυτά για την διατροφή ολόκληρης της περιοχής της Νικαίας. Ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο έφορης γης δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί αυτά είναι γη για τα παιδιά μας, για να επιβιώσουν. Περιμένουμε με προσδο... μεγάλες προσδοκίες τη διαμεσολάβησή σας γιατί για μας πρόκειται για επανειλημμένες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Βόνσης που ομιλεί τόσο αυτόνομα όσο και εξονόμενος εξονόματος του κυρίου Βαλαμπουά. Βαλαμπουά. Αναφερομένο. Και παρακαλώ στο δυνατόν πιο σύντομα. Donc, euh, mesdames et messieurs les députés, chers membres de... Κυρίες και κύριοι βουλευτές και μέλη της Επιτροπής, Ομιλώ εκ μέρου τη οργάνωση ΟΗΕΝ, Πλέν του Βαχ, Κιλαδά του Βαρ. Διαδιάδο του Βαρ. Ο κύριο Βαρόμπο είναι ο πρόεδρο και τον εκπροσωπώ. Θα ήθελα να σα εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η επιχείρηση εθνικού συμφέροντο. αυτή η οργάνωση που ιδρύθηκε το 2008 και που δημιουργήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2007. κάλυπτε την πεδιάδα του ΒΑΡ με στόχο την προστασία των υδάτων και της βιοπικιλότητας. Από τον ποταμό Βάραγκλη το όνομά τη. Ένα ποταμό ο οποίος ε, από ό,τι δείχνουν οι στρατιωτικοί χάρτες πάει από ένα λόφο στον άλλον. Και στη συνέχεια με διευθετήσεις γεών μετατρέπει και σε έφορη για καλλιέργεια Διάδα. Τα νερά είναι πανταχού παρόντα. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες όπως η οδηγία πλαίσιο του 2000 και του 2009 και η εθνική νομοθεσία 2008-2011 που τις μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο πρέπει να τηρηθούν. Πρόκειται για ε, υγρότοπο ιδιαίτερου εθνικού συμφέροντος και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πρέπει να διαφυλαχθούν. 600.000 άτομα τροφοδοτούνται από αυτή την περιοχή ε, σε πόσιμο νερό. Έχει γεωστρατηγική σημασία. Η ε, η δόμηση γίνεται σε περιοχές ε, συλλογής των υδάτων που είναι στην ευρύτερη περιοχή του ΒΑΡ και τις βλέπετε εδώ. Το μικροκλίμα που δημιουργείται από την παρουσία των υδάτων έχει πολύ ε, μεγάλη σημασία για τη βιοπικιλότητα. 261 διαφορετικά είδη καταγράφονται, είδη πανίδας. Διάφορα ε, είδη κυρίως πτηνών, τα οποία σας αναφέρω διεξοδικά στα θελικά. Και αμφίβια, να και οι υπόλοιποι χάρτες. και απαιτείται η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας Natura 2000 για τους προφανείς λόγους παρουσίας όλων αυτών των διαφόρων ειδών. Είχαμε, είχε αποσταλεί μάλιστα μια επιστολή για μια ε, επιχείρηση ανταλλαγής απόψεων και διαβουλεύσεων που αφορά τη τήρηση των αρχών της ε, υπεροχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογίας και την προστασία των πόρων, κοινωνικού μείγματος κτλ. έχουμε πει στην επιστολή σημειώσει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι των πλημμυρών, να ε, κινηθεί αδίποτε πρωτοβουλία για μέτρα στο μέγεθος των ε, αναγκών και εδώ βλέπετε τη συνέπεια στη βιοπικιλότητα γιατί δεν γίνονται σωστά οι μελέτες αντικτύπου όπως εκεί που έγινε μια υποτιθέμενη μελέτη χωρίς κανένα όμως πραγματογνώμονα ε, επιτόπου για την κατασκευή ενός μεγάλου σταδίου και όπου σημειώνουμε πως ε, δεν ελήφθη υπόψη ο κίνδυνος για εξαφάνιση ειδών, όπως άλλωστε αναφέρουμε και στο ΚΑΠ 4000, στη ΣΑΟΓΑ και στις ε, περιοχές όπου συγκλίνουν διαφόροι παραπότομοι του ΒΑΡ. Κίνδυνος ε, δε για εξαφάνιση ακόμη ειδών ή για σπάνιδα ειδών οφειλωμένη στην εξαφάνιση των φυσικών του στροφών λόγω της εξαφάνισης των γεών και γι' αυτό ζητούμε την επαλήθευση των μελετών που υποτίθεται πως έχουν γίνει. 10.000 εκτάρια βλέπετε εδώ, σε πρόβλεψη μόνο. Έτσι λοιπόν η περιβαλλοντική αρχή αναφέρεται σε μια οδηγία πλαίσιο για τις σωρευτικές συνέπειες όπως εδώ βλέπετε από το Σαν Βάχ και από την Γκόντ και παραθέτω ότι σημειώνει πως δεν μπορεί να αξιολογήσει η περιβαλλοντική αρχή τις συνέπειες σε ε, ε, υγροτόπους του Natura 2000 και τις σωρευτικές συνέπειες στην παιδιάδα του ΒΑΡΤ. Η αρμόδια αρχή. Και επίσης, Μα σας παρακαλώ μιλήστε λίγο πιο γρήγορα. Και επίσης καλείται να αναστείλει η αδίποτε χωροταξική δραστηριότητα ώστε να επιτρέψει την περαιτέρω μελέτη των συνεπειών η οποία θα επιτρέψει τον υπολογισμό των συνεπειών δυνάμει και του Natura 2000. Δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις, 22 Σεπτεμβρίου του 2014, με τις συνέπειες, ανάπτυξη, ανάλυση των συνεπειών λεπτομερέστερη για τον συλλογικό ισολογισμό σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, το γεωργικό περιβάλλον, την βιοπικιλότητα, τις ορευτικές συνέπειες ως προς τις μεταφορές που θα πρέπει να αιτιολογηθεί όλος ιδιαιτέρως, συνθετική παρουσίαση ορευτικά των συνεπειών σε μορφή πίνακα και επίσης δεύτερη πρόταση της Δευτέρας Οκτωβρίου στον ίδιο ιστότοπο μάλιστα αναφέρεται που απλώς καταργεί το εν λόγω εδάφιο. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι έπρεπε να έχει γίνει μια οικολογική μελέτη επιπτώσεων που δεν κοινοποιήθηκε ποτέ ούτε στην κοινή γνώμη του στις ε, ενδιαφερόμενες οργανώσεις. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί και καθώς όπως βλέπετε στο χάρτη μας υπάρχει τεράστια επιρροή στην περιοχή μας, με όλα τα ναι, κόκκινα ναι, χρώματα που ναι. έχουμε βάλει στο χάρτη, θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί διεξοδικά. Πρέπει λοιπόν να αναλυθούν τα, καλά, τα, με, τα κατάλληλα μέτρα. Αυτά που είπα τώρα ήταν μόνο για τη συλλογική δράση. Έχω και άλλα όμως να πω. Και θα περάσω στα... Θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο γρήγορα. Θα με καταφέρουν οι διερμηνείς, δεν πειράζει. pouvez être bref si possible. Merci. Aucun problème. Conformément à la pétition de l'association Green que j'ai l'honneur de représenter. Η οργάνωση Green, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, ασχολείται με το δέλτα του εν λόγω ποταμού, παλιά φωτογραφία του 1979 σε ελώδη περιοχή πάνω στην οποία χτίστηκε και το αεροδρόμιο. Εδώ έχουμε κροκάλες και λατίπες έχουμε διάφορα πτηνά, χαρακτηριστικά βλέπετε τις φωτογραφίες εδώ. Ε, έχει χυμαρόδι τύπο και τον, μεγαλύ, τον περισσότερο χυμαρόδι στη Γαλλία ο Βάρα, λόγω της ορεινής του προέλευσης και της παιδινής του κατάληξης και της γεωγραφικής του διαμόρφωσης που επιταχύνει ακόμη περισσότερο τα ύδατά του. Το αεροδρόμιο της Νικαίας είναι χτισμένο πάνω σε ένα γκρεμό ασταθή και σε διαρκή μετακίνηση. η διαρκής ε, δόμηση στην περιοχή του Βάρα οδήγησε στις φωτογραφίες που βλέπετε σε <laughs> πνιγμό το αεροδρόμιο, σε πολυάριθμους θανάτους, καταστροφή της πόλης Αντίμπ. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο πως ε, όσο περισσότερο χτίζεται τόσο χειρότερα είναι τα προβλήματα και οι κίνδυνοι πλημμύρας διάβρωσης των εδαφών και υποβάθμισης των εδαφών. Μάλιστα είχαμε ένα καρφούρ το οποίο έπεσε ο κύριος, το κύριο Θεμέλιο, καταστράφηκε το κύριο Θεμέλιο στήριξη. Το ίδιο αντίστοιχα προβλήματα είχαμε και στο μεγάλο στάδιο. Ήταν εσκεμμένη η α, παραμέληση των ε, μελετών των περιβαλλοντικών, γιατί θεωρήθηκαν υπερβολικά απειλητικές. Εδώ βλέπετε διάφορα είδη πτηνών που κινδυνεύουν από καταστροφή. Υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντολόγοι όπως ο Ζόρς Τεφάρς που παρακολουθούν εδώ και χρόνια τους κινδύνους από την ανθρώπινη δραστηριότητα, απόβλητα μπάρμπεκιου, πικνίκ ε, και άλλη καταστροφική δραστηριότητα. Προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε ότι υπαγόμαστε στην σύμβαση Ράμσαρ για την επέκταση του ΚΑΠ 3.000, ε, ε, μάλλον για το ΚΑΠ 4.000, το καινούριο δηλαδή σχέδιο, θεωρούμε ότι είναι πολύ ευαίσθητη και ευάλωτη περιοχή και ενδυνεύουν ε, ε, ενδιαιτήματα και είδη της Φλωρίδας και της Πανίδας καταστρέφεται ενδιαίτημα σε μεγάλη έκταση και διαταράσσεται λόγω των εργασιών το σύνολο των ε, πτηνών είτε αυτά είναι αποδημητικά είτε όχι. Υπάρχει κίνδυνος οριστικά να εξαφανιστούν τα προστατευόμενα αυτά είδη, κανένα πρόβλημα και σημειώνουμε ότι υπάρχουν σοβαρές παρατηρήσεις σε σχέση με τα ύδατα. Εδώ στο χάρτη που βλέπετε είναι η μορφολογία και η αστάθεια των εδαφών όχι μόνο σε σχέση με τα χαμηλά του ποταμού, αλλά και με τις υψηλότερες ζώνες συλλογής των εδάτων. Καμία ευρωπαϊκή οδηγία δεν έχει υπολογιστεί ή γίνει σεβαστή στο σχέδιο και σε όλες τις προτάσεις που σας εξέθεσα νωρίτερα με την προηγούμενη αναφορά θέλουμε αυτή η προστατευόμενη περιοχή να προστατευτεί πραγματικά, να σταματήσουν τα έργα και τα σχέδια, σχέδια και έργα τα οποία δεν θα έπρεπε καθόλου να έχουν προχωρήσει αφού δεν έχουν γίνει σχετικές μελέτες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των ομάδων, αλλά πρώτα την Κομισιόν. Αλλά να είστε σύντομοι παρακαλώ, ε. Σύντομοι. Ποιος θα μας πει για αυτά από την Κομισιόν. Εγώ κυρία Πρόεδρε. Το ντοσχέ είναι πολύ πολύπλοκο όπως είδατε και εσείς. Υπάρχουν προγράμματα, σχέδια, σχεδιαγράμματα Εδώ πρόκειται για περιφέρεια πολυπληθή και με πολλές πόλεις και λόγω των επιχειρημάτων των αναφερόντων ρωτήσαμε τη Γαλλία μέσω του μηχανισμού EU Pilot για να έχουμε πληροφορίες και η ανάλυση δεν τελείωσε ακόμα, δεν τελείωσε. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία όμως και θα τονίσω μερικά άλλα. Πρώτον, αυτό που λένε οι αναφέροντες αφορά μια συγκεκριμένη οδηγία και θεωρούν ότι ορισμένα σχέδια και προγράμματα που περιέχει έπρεπε να είχαν τύχει προηγούμενης αποτίμηση για τις ε, περιβαλλοντολογικές συνέπειες. Αυτό ακόμα μελετάτε. Αυτό που θα ήθελε να πει η Κομισιόν σήμερα είναι ότι έχει γίνει δίωξη, έχει αρχίσει δίωξη κατά της Γαλλίας ως προς την, ε, ήδη ως προς την μεταφορά της οδηγίας αυτής στο γαλλικό δίκαιο. Καταλαβαίνουμε τη λογική των αναφερόντων, αλλά ούτως ή άλλως εμείς θα ενδιαφερθούμε μάλλον στο διαρθρωτικό πλάι πρόγραμμα. Τώρα για την αποτίμηση των συνολικών αποτελεσμάτων ούτε αυτή η αποτίμηση δεν έχει τελειώσει και ως προς τα υπόλοιπα την οδηγία για τα ύδατα δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που λάβαμε από τις γαλλικές αρχές, δεν θεωρούμε ότι δικαιολογείται εδώ να θεωρηθεί ότι έγινε παραβίαση κοινοτικού δικαίου. Για τα πιο, προχωρη, πιο προχωρημένες φάσεις του σχεδίου έχει γίνει αποτίμηση και δεν βλέπουμε καμία παραβίαση. Τώρα για την φύση. Οι γαλλικές αρχές έλαβαν υπόψη τους τις αποτιμήσεις και πάλι δεν αποδεικνύεται πουθενά παραβίαση. Ιδίως για την οδηγία των βιοτόπων. Όσο για τις πλημμύρες, για μας Αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στην αποτίμηση που έχουμε. Και τέλος, θα ήθελα να σας τονίσω το ότι οι αναφέροντες έχουν κάνει προσφυγή εθνικά για το πώς. Πώς. Και συγκεκριμένα για τις πλημμύρες θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο εθνικός δικαστής δικάζει και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και εκείνος θα κρίνει επί τόπου τι συμβαίνει και όχι εδώ εμείς από την Κομισιόν. Μάλιστα. Λόγος τώρα στην κυρία Ριβαζή να ευχαριστήσω όλες τις οργανώσεις που είναι εδώ παρούσες γιατί έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και εγώ σαν βουλευτής θα ήθελα να μιλήσω για την εκλογική μου περιφέρεια κατά κάποιο τρόπο στην οποία έχω πάει επανειλημμένα και να σας μιλήσω λίγο για το κλίμα. Δεν βρισκόμαστε οπουδήποτε. Ε. Βρισκόμαστε στην πεδιάδα του ΒΑΡ που υπάρχει η, νίκη, η Νίκαια, η πόλη της Νίκαιας και υπάρχει και ένα πολιτικό κλίμα πολύ δύσκολο. Και ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου προφανές να έχουμε τέτοιου είδους οργανώσεις σε επίπεδο δημοκρατίας. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση. Οι δημόσιες αυτές διαβουλεύσεις ζητήθηκαν, υπήρξαν τέσσερις σε μικρούς χώρους, υπήρξε και μία στην Νίκαια. Και πράγματι υπάρχει όμως μια έλλειψη δημοκρατίας και χρειάστηκε να πιέσουμε πολύ έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική συζήτηση. Δεύτερον, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω στα πλαίσια αυτού του κλίματος το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται διότι πολιτικά και εκεί έχουμε ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητάμε ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά του Προέδρου της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Περιοχής ασκούνται πιέσεις ε, και προς τη δικαιοσύνη γιατί όταν ε, λένε προς τη δικαιοσύνη πήρατε κάποιες αποφάσεις αρνητικές αυτές δεν χρειάζεται και να τις συμπεριλάβετε στη νέα σας απόφαση. Ασκείται λοιπόν μια πάρα πολύ ισχυρή πίεση προς τη ΣΜΚΙΟ. Μετά μας λέτε ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις σε σχέση με τους υδάτινους πόρους. Δεν ξέρω αν το είπανε επαρκώς ε, η ΜΚΟ. Ο, ο κύριος ε, Εστροζή, ο περιφερειακός πρόεδρος δηλαδή, θέλει να κάνει υποτίθεται ε, μια οικοκυλάδα. Και τι θα υπάρχει μέσα στην οικοκυλάδα, την πράσινη κοιλάδα του Εστροζή, τσιμέντο. Θυμηθείτε τι έγινε στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου. Μέσα σε ελάχιστες μέρες έπεσε πάρα πολύ νερό, διότι συμβαίνει και αυτό αλλά με τον τεχνητό τρόπο με τον οποίο αντικαθιστούμε τα εδάφη δημιουργούμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε το Παγκόσμιο Κέντρο για την Επιχειρηματικότητα. Έχουμε την πολυτροπική ε, ε, ε, έδρα του πολιτιστικού κέντρου. Έχουμε επίσης και ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο, ένα πολυτροπικό σταθμό μεταφορών θέλουμε να μεγαλώσει το αεροδρόμιο. Και εκεί ε, που υπάρχει και η υπάρχουσα αγορά θέλουμε να τη μετακινήσουμε για να χτίσουμε ακόμα περισσότερο, να γκρεμίσουμε το στάδιο. Έχουμε την παρόν Αγκοστιέρ, ε, μια μεγάλη αγορά αγροτικών προϊόντων, την οποία και αυτή θέλουμε να συμμετώσουμε. Ε, πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά και τι η κοκκιλάδα είναι αυτή αν εσείς συνεχίσετε να τσιμεντώνετε τις αγροτικές περιοχές. Η απάντηση είναι ότι σε επίπεδο ε, φύσης ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, στο δέλτα του Βαρ υπάρχει μια τεράστια ζώνη με μεταναστευτικά πουλιά. Στα πλαίσια του ΚΑΠ 3000 θέλουμε να μεγαλώσουμε τις βιομηχανικές ζώνες και δημιουργώντας και υπόγεια πάρκινγκ. Ε, από τις Κάνες, το Μοντελιό και το Σαν του Βάρ υπήρξαν 20 νεκροί. Και πού πνίγηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα υπόγεια πάρκινγκ. Θέλουμε λοιπόν να τσιμεντώσουμε ακόμα και καταλαβαίνετε ε, ο Βάρ δεν είναι ένας ήρεμος δόν, είναι πραγματικά ένας χυμαρόδης ποταμός. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο και τις ε, οδηγίες σας σε σχέση με τους συνδυασμούς των επιπτώσεων. Η περιφέρεια αρνήθηκε να δώσει θετική γνώμη. Η Αντρεάλ που είναι οι υπεύθυνε περιβαλλοντικές αρχές είπαν ότι δεν συμφωνούν καθόλου με την τροποποίηση της περιοχής του Σεν Λορόντιβάρ και της Γκόντ και ζητούν τις πιθανές διασταυρούμενες επιπτώσεις. Υπάρχουν επιμέρους πάρα πολλά σαλαμοποιημένα προγράμματα και δεν υπάρχει καμία συνολική πρόταση. Δεν υπάρχει σεβασμός των οδηγιών. Λέτε ότι όταν βλέπετε τα λεγόμενα οικολογικά, ή τις οικολογικές περιφέρειες των πόλεων, δεν είναι τίποτα, αυτά είναι λόγια θα πρέπει οι γαλλικοί νόμοι να γίνουν σεβαστοί. Και ε, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί αλλά όχι με τέτοιου είδους επιμέρους προτάσεις. Έχω πάει επανειλημμένα, έχω συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή του προγράμματος και κατάλαβα από πλευρά του ότι αν δεν βοηθηθεί εκ των άνω δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την απειλή. Υπάρχει λοιπόν μια άσκηση πίεση τρομακτική εις βάρος αυτού του εδάφους. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε. Μάρτεν. Εγώ θα είμαι σύντομος πρόεδρε. Μην ξανακάνουμε τέτοια συνεδρίαση. Να περάσουμε τους αναφέροντες στο τέλος ενώ μπορεί να έχουν αεροδρόμια, τρένα κτλ. Στοιχειώδης ευγένεια θα απαιτούσε να τους ακούσουμε πρώτους. Αυτό το λέω τυπικά τώρα. Και τους πιέζουμε και αναγκάζονται να μιλήσουν πιο γρήγορα εκεί δυσκολεύονται οι διερμηνείς τέλο πάντων. Επί της ουσίας τώρα, ευχαριστώ τους αναφέροντες που ήταν τόσο σαφείς, σαφέστατοι. Αλλά τι συζήτηση να γίνει εδώ πέρα, υπάρχει το δίκαιο, αλλά υπάρχει και η κοινή λογική. Και βλέποντας αυτά που είδαμε, τους αριθμούς, δεν χρειάζεται να είναι κανείς εμπειρογνώμων για να καταλάβει ότι πρόκειται για υπερβολές, ιδίως μερικές εβδομάδες μετά τις καταστροφές των πλημμυρών με πάνω από 20 νεκρούς σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να κρατήσει φυσικά ανοιχτή την αναφορά, να γίνει μια γενικότερη μελέτη επιπτώσεων πέρα από τα συγκεκριμένα τα πουλάκια, τα νερά και τα λοιπά, κάτι πιο σφαιρικό και όχι με σαλαμοποίηση. Για να θυμηθούμε και εμείς και η Κομισιόν ότι χθες μόλις ψηφίσαμε μια έκθεση προηδείας πρωτοβουλίας πολύ σημαντική για την COP21 που θα οργανωθεί όπως ξέρετε στη Γαλλία. Καλό είναι να ζητάμε την καταπολέμηση των εκπομπών διοξιδίου, αλλά επίσης καλό είναι να σεβόμαστε και να διατηρούμε το φυσικό περιβάλλον, γιατί και αυτό θα βοηθήσει. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι αξιοθρύνητο να συνεχίζεται η τσιμέντωση. Το είπε και η κυρία Ριβαζή, σε μια περιφέρεια μάλιστα που είναι ήδη πολύ πυκνοκατοικημένη να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να γίνει μια γενική μελέτη επιπτώσεων. Αντικτύπου. Ευχαριστούμε κύριε Μαρτέν μου. Κύριε Λαφριγέ. Ναι κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια. Εγώ σημερίζομαι ένα τμήμα, ίσως και όλα, αλλά κυρίως ένα τμήμα αυτών που είπαν οι αναφέροντες αλλά θα ήθελα να μας στείλουν ιδίω τους Γάλλους βουλευτές όλα τα έγγραφα που μας παρουσίασαν. Ξέρω ότι βιάστηκαν και χρειάστηκε να μιλήσουν πολύ γρήγορα αλλά ακόμα και ως γαλλόφωνος mm. γηγενής δεν τα κατάλαβα όλα Φαντάζομαι λοιπόν όσοι ξέρουν λιγότερα καλά γαλλικά από μένα τι πρόβλημα αντιμετώπισαν οι μεταφραστέ ιδίω. Γιατί η παρουσίαση έγινε υπερβολικά γρήγορα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω και εγώ αυτό το φάκελο τα έγγραφα για να καταλάβω. Και όταν τα καταλάβω τότε θα εκφραστώ και εγώ πιο σαφώς. Παρ' όλα αυτά. Ακούω ότι μας λέει και η Κομισιόν, χωρίς να υπησέλθω στην ουσία. Μας λέει ότι κατά αυτήν δεν υπήρξαν παραβιάσεις του δικαίου και αν υπάρξουν, εφόσον έχουν μεταφερθεί στο γαλλικό δίκαιο, πρέπει να γίνει προσφυγή σε γαλλικό δικαστήριο. Άκουσα επίσης την κυρία του αν δεν απατώμε να λέει ότι υπάρχει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί εκδοθεί απόφαση. Επομένως πώς να εκφραστούμε όταν δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όλες οι δυνατές εθνικές προσφυγές. Αυτός είναι συνήθως ο κανόνας για τις αναφορές. Γιατί εμείς δεν κάνουμε μια ποιοτική αξιολόγηση εδώ πέρα, ό,τι θέση να έχουμε. Είναι να παληθεύουμε ότι ο πολίτης δεν αντιμετωπίζει έναν τείχο και αλλά αφού έχει εξαντλήσει όλες τις ένομες οδούς. Αλλά εφόσον υπάρχει προσφυγή, επειδή έχω εμπιστοσύνη απριόρι στη δικαιοσύνη της χώρας μου, θα ήθελα να περιμένουμε να δούμε τι θα πει αυτό το δικαστήριο. Yeah nous serons amenés à, à nous revoir très θα τα ξαναπούμε αναγκαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πάρετε κι εσείς ξανά το λόγο κυρία του Ζώμου. Ναι, ένα λεπτάκι για να πω στον κύριο αυτόν ότι θα στείλουμε πλήρες, πλήρη φάκελο η προσφυγή μόλις κατατέθηκε για να ζητήσουμε το λόγο από το γαλλικό κράτος. Αλλά για το πέσο όχι το πώς κυρία μου. Εννοώ ότι όπως είπε και η κυρία Λεβαζή υπάρχουν ισχυρές πιέσεις και οι επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται εθνικού ενδιαφέροντος ενώ εμείς βλέπουμε ότι η μεταφορά του μην γίνεται μόνο και μόνο για να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο που ενδιαφέρει τον Δήμαρχο. Για μας το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη απαρχαιωμένο γίνεται μια επένδυση για μια απατηλή ανάπτυξη, δίθεν ανάπτυξη σε ζώνη που μπορεί να πλημμυρίσει εύκολα. Και παρόλα αυτά ο Δήμαρχος λέει ότι σέβεται το δίκαιο. Χρειαζόμαστε τη μεσολάβησή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τους μεν και τους δεν και τώρα που ακούσαμε και τους βουλευτάς μπορούμε να καταλήξουμε λέγοντας ότι θα κρατήσουμε την αναφορά αυτή, αυτές τις αναφορές ανοιχτές και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας της Κομισιόν. Τα ακούσαμε όλα λοιπόν και θα περιμείνουμε, το ξαναλέω, την απάντηση της Κομισιόν. Και τότε θα μπορέσουμε να πούμε τι θα κάνουμε. Τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης, ακόμη μία αναφορά ισπανική για τους εμπορικούς φραγμούς στην πόλη Μπέγκες στην Ισπανία. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ρεδόνδο. Ε, δεν θα ήθελα να δείξω ότι είμαι αγενής απέναντι στους Ισπανούς φίλους σήμερα και δεν ήρθα να κάτσω μόνο για τους Γάλλους, θα ήθελα όμως να κάτσω και για τους Ισπανούς αλλά δυστυχώς πρέπει να γυρίσω στην περιφέρειά μου και θα ήθελα στα πλαίσια της γνωστής γαλατικής ευγένειας να ζητήσω συγγνώμη για την αποχώρησή μου, υποχρεωτική αποχώρηση. Η κυρία Ρεντόντο. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ όλους. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Ρεντόντο. Το Μπέγες είναι στην περιφέρεια της Μαρκελόνης από το 2009 δημιουργήθηκε μια νέα διαχειριστική δημοτική αρχή ο οποίος ε, καθορίζει τα διαφορετικά επίπεδα εμπορευματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχει υπάρξει από τότε μια μείωση των ε, επιχειρηματικών και εμπορικών ε, καταστημάτων και η κεντρική περιοχή της πόλης δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές ε, ε, ανάγκες και δεν ενισχύεται η επιχειρηματικότητα. Χρησιμοποιείται με πολύ περιοριστικό τρόπο η αδειοδότηση, το μέσο της αδειοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έγινε είναι να περιοριστεί η αύξηση των εμπορικών καταστημάτων και αυτό είναι κάτι το οποίο επηρέασε τον δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής εις βάρος της απασχόλησης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες λοιπόν. Οι πολιτικές ρύθμισης όλων αυτών των εμπορικών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να ε, υποβάλλονται πλέον σε τόσες περιοριστικές διατάξεις. Η οδηγία για τις υπηρεσίες καθορίζει την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ο Ισπανικός νόμος προβλέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε εμπορικές δραστηριότητες. Είναι συμβατή με την εμπορική ε, ε, με την κοινοτική ρύθμιση, την κοινοτική οδηγία και δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε και να επιβάλλουμε ποσοτικούς και εδαφικούς περιορισμούς με όρια τα οποία καθορίζονται ε, μόνο με τον αριθμό του τοπικού πληθυσμού. Η συγκεκριμένη αυτή απόφαση περιορίζει τον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων. Επίσης περιορίζει και τον αριθμό των εστιατορίων κτλ. Η τοπική κυβέρνηση συνειδητοποιούν, συνειδητοποιεί τη δυσκολία του προβλήματος αλλά δεν έχει αποκαταστήσει την ευρωπαϊκή τάξη. Η νομική υπηρεσία του Δήμου εξέδωσε στις 5 ε, Οκτωβρίου του 2010 ε, το έχουμε καταθέσει, την έχουμε καταθέσει την έκθεση αυτή λέγεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση αυτή του Δήμου είναι αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Ισπανική νομική ρύθμιση. Και θα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση αυτή με βάση την ομοφωνία ή τη μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης των Βέουες. Κάτι τέτοιο δεν θα επέτρεπε τον περιορισμό των δραστηριοτήτων και των εμπορικών υπηρεσιών. Ε, το Φέγας λοιπόν, με, το οποίο είναι μια εμπορική πόλη με έναν αρκετά σημαντικό αριθμό του πληθυσμού, ε, αναγκάζει τους πολίτες της να πηγαίνουν σε γειτονικές πόλεις και εγκαταστάσεις για τραπεζικές δραστηριότητες ή άλλες αγοραστικές δυνατότητες. Γι' αυτά όλα λοιπόν ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρώτον να αναζητήσει τα στοιχεία της καταγγελίας μας, σαν δεύτερον η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση σε σχέση με την αξιολόγηση του Δημοτικού Διατάγματος το οποίο ρυθμίζει τις εμπαρικές δραστηριότητες στην επαρχία της Βαρκελόνης, στην πόλη της Μπέγουετς και να δει σε ποιο βαθμό είναι συμβατές οι ρυθμίσεις αυτές με την κοινοτική οδηγία και με τον Ισπανικό νόμο 1798 της 23ης ε, Νοεμβρίου σε σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες ε, ε, παροχής υπηρεσιών. να δούμε σε ποιο βαθμό είναι αντίθετες οι ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται με το νόμο στο άρθρο 11 και στο άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες που λέγεται ότι ο διακανονισμός και η ρύθμιση της πρόσβασης σε εμπορικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να υφίσταται εδαφικές ή ποσοτικές πιέσεις περιορισμού με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός του πληθυσμού ή ο αριθμός των εμπόρων και είδαμε τι συνέπειες έχει η ερμηνεία αυτή, η εφαρμογή μάλλον αυτή της ερμηνείας σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Είναι αντίθετη και με την οδηγία, είναι αντίθετη και με τον νόμο 17 ε, του Ισπανικού κράτους συμπερασματικά. Εάν πράγματι η οδηγία λέγει ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού εδάφους, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που δημιουργούν προβλήματα σε μια πολύ δυναμική αγορά που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στους περιορισμούς χρήσης του κέντρου της πόλης της Βέγουας και θα πρέπει αντίθετα να διευκολύνουμε την ελευθερία εγκατάστασης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και σύμφωνα και με, τις, με το τρίτο άρθρο 144 του Ευρωπαϊκού και του Ισπανικού νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα την αναφορά και θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες σέβεται μεν την ελευθερία εγκατάσταση αλλά θέλει να υπάρξουν περιορισμοί μόνο αν υπάρχει λόγος γενικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή το γενικό ενδιαφέρον είναι κάτι χωροταξικό. Κατανοώ το παράπονο των αναφερόντων, αλλά υπάρχει η απόφαση του Δήμου του Μπέγκουες και από που φαίνεται ότι ο στόχος είναι η εξισορρόπηση μεταξύ εμπορικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων υπηρεσιών. Αναρωτιόμαστε λοιπόν και ρωτήσαμε ήδη από τους αναφέροντες, ζητήσαμε παραπάνω πληροφορίες, αναρωτιόμαστε πώς μπορεί μια τέτοια διευθέτηση να οδηγήσει σε μείωση των εμπορικών καταστημάτων. Ο στόχος φαίνεται να είναι μάλλον η καλύτερη διοργάνωσή τους και όχι ο περιορισμός τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, διαβάζοντας την απόφαση του Δήμου δεν βρήκαμε αυτά που κατηγορεί αναφέρουσα, δηλαδή την, την ελάχιστο, την ελάχιστη απόσταση την οποία αναφέρει ή την πυκνότητα των εμπορικών καταστημάτων όπως είπε δύο τράπεζες ανά δρόμο. Αν μου επιτρέπετε δεν θα ήθελα να προσθέσω ότι στο προήμιο αυτής της απόφασης του Δήμου υπενθυμίζεται ότι μπορεί να προσφύγει κανείς στο τοπικό δικαστήριο της περιφέρειας εκείνης απευθυνθήκατε εκεί. Όπως είπε η συνάδελφος για την προηγούμενη περίπτωση, ο πρώτος αρμόδιος δικαστής είναι ο τοπικός, ο περιφερειακός, που μας φαίνεται το καλύτερο επίπεδο για να απευθυνθείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα μέλη. Ευχαριστώ. Θέλω να καλωσορίσω. Ευχαριστώ. Θέλω να καλωσορίσω τους αναφερομένους και θέλω να ευχαριστήσω και για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι τίθεται θέμα εδώ σε σχέση με το σεβασμό της οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι προβλέπεται σαφώς και το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις στην περίπτωση κατά την οποία τίθενται θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας. Το θέμα είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις υπηρεσίες και στις εμπαρικές δραστηριότητες και δεν ξέρω εδώ τι αμφιβολίες θα μπορούσα να είχα σε σχέση με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με την αναφορά. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο, διαφορετικές, ε, με δύο διαφορετικούς ισχυρισμούς. Είναι σαφές ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για να διαμορφώσουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη. Θα πρέπει να παραμείνει λοιπόν ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά να συλλεγούν από όλε τις πλευρές περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες έτσι ώστε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο στην ουσία παρουσιάζεται σαν ένας περιορισμός των δραστηριοτήτων των εμπορικών, κάτι το οποίο εμάς σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μας ενοχλεί. Ε, ε, I think... Το... Θα συμφωνήσω, θα χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες. Ας μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά για να δούμε και την αξιολόγηση της Επιτροπής και περαιτέρω τι μπορεί να γίνει. Καλή ιδέα λοιπόν. Αλλά πριν κλείσω τη συνεδρίαση, οι αναφερόμενοι έχουν κάτι επιπλέον να πούν. Ποιος θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. La representante de la Comisión Europea eh, alude objetivos de interés general Πράγματι υπάρχουν ορισμένοι γενικοί στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί σε σχέση με τις ρυθμίσεις της χωροταξικές. Αυτή δεν είναι η άποψη των πολιτών συγκεκριμένα της πόλης μας. Έχουμε προβλήματα σε σχέση με τον ορισμό των υπηρεσιών ας πούμε που παρέχονται. Καταλαβαίνει κανείς ότι για να μπορέσει να πάει σε ένα γιατρό το απόγευμα σαν παράδειγμα θα πρέπει να πάει σε μια περιοχή 11 χιλιόμετρα πιο, 8 χιλιόμετρα πιο μακριά και δεν υπάρχει δεύτερο φαρμακείο, δεν επιτρέπεται να, και θα πρέπει να χρειαστεί να πάρουμε το αυτοκίνητο και να πάμε επίσης 8 χιλιόμετρα πιο μακριά. Υπάρχουν περιορισμοί λοιπόν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες Στην ουσία το πρόβλημα αυτό επανέρχεται και τίθεται με διαφορετικό τρόπο από όλες τις πλευρές. Και Por ejemplo, dice que no hay λέει σαν παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με τις επιφάνειες των εμπορικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό δεν είναι αλήθεια στις τράπεζες σαν παράδειγμα απαιτείται να είναι 12 μέτρα η μία πιο μακριά από την άλλη. Και επίσης υπάρχουν θέματα και με τις δευτερεύουσες εξόδους των διαφόρων κτηρίων που είναι απαραίτητες για να πάρουν άδειες εκμετάλλευσης. και αν οι αποστάσεις αυτές είναι μικρότερες των 12 και φτάνουν μέχρι τα 11 τότε καταλαβαίνετε ότι λειτουργούν σωρευτικά οι περιορισμοί αυτοί και δεν μπορεί να ανοίξει ένα μπαρ στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν γενικότερα προβλήματα ερμηνείας σαν παράδειγμα. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει και μια παραανάγνωση θα έλεγα των προβλημάτων. Ακούστηκε ότι μπορεί να μην υπάρχουν πάνω από δύο τράπεζες στον ίδιο δρόμο. Όχι δύο τράπεζες στον ίδιο δρόμο, δύο τράπεζες στο σύνολο της περιοχής, του κέντρου της πόλης των Βέγας. Δεν ξέρω λοιπόν αν πραγματικά οι στόχοι της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης ε, στην οποία προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η ισορροπία. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα λέγει ότι ο νόμος 17 του 2009 σύμφωνα με τον ίδιο Γενικό Γραμματέα δίνει διαφορετικές δυνατότητες σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Λοιπόν, τελειώνοντας μια σκέψη. Ένα, μια απόφαση του Δημοτικού Συμφουλίου λοιπόν κρίνεται ουσιαστικά από την κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βοηθάει την ευημερία του λαού, να βοηθάει την οικονομία, να βοηθάει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη, κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη απόφαση αυτή, η οποία δεν διευκολύνει την οικονομική ευημερία της πόλης των Μπέγουες. Για μια πόλη μιλάμε η οποία κυρίως ζει από τις υπηρεσίες και από τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. πολύ. Όπως είπαμε, είναι ανοιχτή αναφορά μέχρι να λάβουμε τις πληροφορίες. για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στο σύνολό τη. Ολοκληρώνουμε τι εργασίε μα. Ευχαριστώ τους συναδέλφου, γραμματεία, διερμηνείς λέει ο Πρόεδρος. Καλό βράδυ.